staatspräsident Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Πλεβέινα, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μεγάλη τιμή η παρουσία σας εδώ σήμερα. Για πολλά χρόνια ήσασταν σε στενή επαφή ως πρόεδρος της χώρας σας, που είναι σημαντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλατε στις στενές σχέσεις. Και εδώ και δύο χρόνια αντιμετωπίζουμε από κοινού την πρόκληση της ε, μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψή σας. Κύριε Πρόεδρε Πλευνέιεφ, είναι τιμή μας που είστε ε, εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξοχότητες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, είναι προνόμιο πραγματικά που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα και απευθύνομαι σε εσά ως πρόεδρος της Βουλγαρίας. Πραγματική τιμή να μπορώ να μιλάω εδώ, στην πραγματική καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Είμαι ένας περήφανος φιλοευρωπαίος πρόεδρος ενός φιλοευρωπαϊκού έθνους. Εμείς οι Βούλγαροι είμαστε περήφανοι που μπορούμε να αποτελούμε παράγοντα σταθερότητας και θετικών εξελίξεων στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι κοινό μας καθήκον να περασπίσουμε τις αξίες ευρωπαϊκές όσον αφορά την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την αλληλεγγύη. Και Κοινό μα στόχο να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε την ιστορία στα πλαίσια ενός σχεδίου για μια ενωμένη και ειρηνική Ευρώπη. Η ειρήνη όμως και η ελευθερία δοκιμάζονται σήμερα και δέχονται επιθέσεις. Αντιμετωπίζουμε σήμερα τη χειρότερη κατάσταση ως προς την ασφάλεια από τότε που τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Βρίσκουμε θεμελιώδεις διαφορές αυτή τη στιγμή μεταξύ παγκοσμίων και περιφερειακών δυνάμεων. Τα εθνικά σύνορα και οι διεθνεί αρχέ αυτή τη στιγμή τίθενται ένα αμφιβόλο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύπλοκο διεθνέ σύστημα όπου παγκόσμιοι και περιφερειακοί θεσμοί και δυνάμει αδυνατούν πλέον να αποτρέψουν αλλά και να επιλύσουν τον πρωτόγνωρο αριθμό συγκρούσεων που γνωρίζουμε σήμερα. Σε πολλέ περιοχέ ο πόλεμο και ο τρόμος επικρατούν. Τα κράτη και οι θυσμοί διαλύονται. Σήμερα λοιπόν στην Ευρώπη συνειδητοποιούμε ότι οτιδήποτε συμβαίνει στη Μέση Ανατολή ή στην Αφρική επηρεάζει και τις ζωές μας εδώ άμεσα. Βλέπουμε ότι επί του παρόντος επανέρχονται τα σύνορα. Ότι η γενιά εκείνη η οποία έριξε το τείχος του Βερολίνου είναι η ίδια που οικοδομεί νέα τείχη στην καρδιά της Ευρώπης. Ναι, όντως, επικρατεί ανισορροπία στο σημερινό κόσμο και θα πετηθεί χρόνο προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια νέα ισορροπία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ασταθεί περιοχέ, μια ασφαλή σύνορα και πολίτε οι οποίοι ανησυχούν. Η τρομοκρατία αναδύεται. Οποιαδήποτε στιγμή, ανα πάσα στιγμή, μπορεί να συμβεί με τρομοκρατική επίθεση. Κανεί δεν είναι ασφαλή. Σήμερα λοιπόν η εξουσία στο σημερινό κόσμο μετατοπίζεται και παίρνει άλλες μορφές. Στη διάσκεψη για την ασφάλεια που έλαβε χώρα στο Μόναχο, ο Ρώσος Πρωθυπουργό μίλησε για την περίοδο του πρώτου ψυχρού πολέμου και για την εποχή του νέου ψυχρού πολέμου που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ελπίζω ότι δεν οδεύουμε προς ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Δεν διανύουμε μια περίοδο νέου ψυχρού πολέμου, αλλά μάλλον βρισκόμαστε σε μια περίοδο ψυχρής ειρήνης. Πριν από δύο χρόνια, στη διάσκεψη για την ασφάλεια του Μονάχου, Είχα τονίσει ότι η Ευρώπη έχει περάσει πλέον σε μια νέα περίοδο. Η Ουκρανική κρίση άλλαξε τα δεδομένα. Έχουμε περάσει λοιπόν σε μια νέα φάση ανάπτυξης, την οποία εγώ αποκαλώ περίοδος ψυχρής ειρήνης. Ειρήνης μεν, γιατί ουδής επιθυμεί τον πόλεμο, αλλά ψυχρής ειρήνης από την άλλη, γιατί βλέπουμε αντιπαραθέσεις και μεθόδους από την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Πόλεμοι προπαγάνδας, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, πόλεμοι δια αντιπροσώπων, Πόλεμη προπαγάνδας και ορισμένες χώρες ψυχράθηκαν, αποσταθεροποιήθηκαν και αποδυναμώθηκαν μέσω των παγωμένων συγκρούσεων. Ο Ρώσος Πρόεδρος πολύ συχνά αναφέρεται σε μια νέα ισορροπία σε έναν κόσμο με νέες σφαίρες συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων. Οδεύουμε πραγματικά προς μια νέα διάσκεψη της Γιάλτας. Αν το επιτρέψει αυτό η Δύση, τότε αυτό θα αποτελέσει πραγματικά ιστορικό όνειδος. Θα πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα θα πρέπει να προασπιστούμε το δικό μας το όραμα, το δικό μας το όραμα για τη δική μας την ενωμένη την Ευρώπη. Διανύουμε δύσκολες εποχές γιατί οι παγκόσμιοι και περιφερειακοί ηγέτες δείχνουν διαφορετικέ προσεγγίσει και διαφορετικού στόχου όσον αφορά την πολιτική που ακολουθούν. Στόχο ευφυού πολιτική είναι να εξυγχρονίσει, να εκπαιδεύσει, να προωθήσει τη διπλωματία και όχι τον πόλεμο. Αν όμω δεν έχει κανεί συγκεκριμένου στόχου και σκοπού, τότε καταλήγει στον πόλεμο. Χρειάζεται έναν βολικό και εύκολο εχθρό. Είναι εύκολο να αποσταθεροποιεί κανεί. Ολόκληρα κράτη μπορούν πάρα πολύ εύκολα να διαλυθούν από ισχυρού γείτονε. Αλλά οι διαλυμένε κοινωνίε μπορούν να αποκατασταθούν μόνο μέσω των λαών και των ανθρώπων και όχι από τι μεγάλε δυνάμει. Πολύ εύκολα και γρήγορα μπορεί να καταστρέψει κανείς την τάξη, αλλά απαιτείται πάρα πολλή χρόνος για να ανοικοδομήσει κανείς και δυστυχώς αυτό βλέπω σήμερα σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης. Ο στόχος λοιπόν μιας ευφυού πολιτικής δεν θα πρέπει να δημιουργεί περαιτέρω παγωμένες συγκρούσεις και να εισβάλλει στο έδαφος γειτονικών χωρών. Στον 20ο πλέον πρώτο αιώνα δεν είναι φιές να μετακινεί κανείς τα σύνορα, αλλά θα πρέπει να σκέφτεται κανείς πέρα από τα σύνορα. Στόχος μιας ευφύου πολιτικής λοιπόν θα είναι τα έθνη να είναι όσο καλύτερα γίνεται εκπαιδευμένα, ευήμερα, να δυναμώνονται οι πολίτε και να ζουν σε ελεύθερες και ανεκτικές κοινωνίες. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στην εποχή των μεγάλων δυνάμεων, την εποχή εκείνη που χώριζαν μεταξύ τους τις σφαίρε επιρροή του. Δεν μπορούμε για άλλη μια φορά να επιτρέψουμε στα πολιτικά συμφέροντα να διχάσουν τα κυρίαρχα κράτη ή να απειλήσουν την ακαιρεότητά του. Τα όσα συνέβησαν στην Ουκρανία αποτελούν επικρή υπενθύμηση ότι τα επιτεύγματα τη ανθρωπότητα δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Ουδέποτε θελήσαμε έναν πόλεμο πάλι στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώ σήμερα έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη και αυτό βρίσκεται στην Ουκρανία. Για μένα, για μα, η Κρυμαία είναι Ουκρανία και η Ουκρανία είναι Ευρώπη. Και θεωρώ ότι η άρση της υποχρέωσης θεωρήσεων για τους πολίτες Ουκρανίας είναι επιτακτική ανάγκη προκειμένου να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και προκειμένου οι πολίτες της να υποστηριχθούν όπως πρέπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωπαίους. Το δεν γνωρίζουμε πολύ σωστά το παρελθόν πολλές φορές, το δεν έχουμε αντλήσει διδάγματα από την ιστορία, δυστυχώς συνεχίζει και επισκιάζει το μέλλον μας. Δεν θα πρέπει να δώσουμε καμία ευκαιρία στους λαϊκιστές να εκμεταλλευτούν την άγνοια και τη λύθη και να αλλάζουν το παρελθόν κατά το δοκούν. Χαιρετίζω λοιπόν τη δημιουργία του σπιτιού της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η μνήμη του τραγικού παρελθόντος θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να μεταλαμπαδεύεται στις νέες γενναίες. Και αυτό το οποίο πρέπει να περάσουμε προς τις νέες αυτές γενναίες και το πιο σημαντικό μάθημα θα έλεγα, είναι ότι δεν είναι δεδομένη η ειρήνη και ότι αναπόκειται στον καθένα μας να την προστατεύσει. Και ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία πολέμου. Η ειρήνη σημαίνει ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου. Κάθε νέος, κάθε νέος Ευρωπαίος θα πρέπει να είναι σε θέση να δει πόσα και γιατί έλαβαν χώρες όπως η χώρα του Βερντάνη της Λοϊράνης, και για ποιο λόγο δεν θα πρέπει να καταλήξουμε εκ νέου στον πόλεμο. Ο Βούλγαρος επαναστάτης Γκότσε Ντέλτσεπ ονειρευόταν με το μελλοντικό κόσμο που τα έθνη θα κατέληγαν ποτέ πάλι στο πεδίο της μάχης, όπου τα έθνη θα συναγωνίζονταν μόνο στον τομέα του πολιτισμού, της επιστήμης και της γνώσης. Στον 20ο λοιπόν πρώτο αιώνα οι διαφορές της Ευρώπης θα πρέπει να επιλύονται στα κοινοβούλια και όχι στα πεδία μάχης. Η ευρωπαϊκή λοιπόν ολοκλήρωση, το σχέδιο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ακριβώ αυτό το όνειρο προσπαθεί να το κάνει πραγματικότητα. Βέβαια, η Ευρώπη δεν μπορεί να αποτελέσει νησίδα σταθερότητα σε έναν ωκεανό παγκόσμια αστάθεια σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανή αριθμό κρίσεων. Επιπλέον κρίσει διαφαίνονται στον ορίζοντα. Για παράδειγμα, ένα πιθανό Brexit. Η άνοδο εθνικιστών και λαϊκιστών, η μετανάστευση και άλλε κρίσει δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην Ευρώπη να βυθιστεί σε μια ηθική κρίση. Μια κρίση έλλειψη αλληλεγγύη, μια κρίση αξιών. είτε μιλάμε για την μετανάστευση ή για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. Μία οικογένεια είμαστε και οι οικογένειες παραμένουν ενωμένε όταν διανύουν κρίσεις. Και κάθε μέλος της οικογένειας αυτής θα πρέπει να συμβάλλει για την επίλυση και όχι για την όξυνση των προβλημάτων. Η Βουλγαρία είναι περήφανη που ανέκαθεν ήταν μέρος της ευρωπαϊκής λύσης και δρά με τρόπο αλληλέγγυο και υπεύθυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερη σημασία και ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση λόγω των ειρηνικών συζητήσεων και της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών, λόγω των κοινών θεμελιωδών δικαιωμάτων και κανόνων και λόγω του πρωτοφανούς επίπεδου συνεργασίας μεταξύ των 28 κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μοναδικό σχέδιο για την ειρήνη, όπου κάθε έθνος είναι σημαντικό. Κανένα κράτος δεν θεωρείται δευτερεύον ή υποδέστερο. Τα προβλήματα της μετανάστευσης, τρομοκρατίας, κλιματικής αλλαγής, οικονομικής κρίσης και άλλα υπερβαίνουν τα σύνορά μας. Τα προβλήματα αυτά είναι διεθνικά και απαιτούν κοινέ προσπάθειες. Η συνεργασία δεν αποτελεί πλέον απλή επιλογή, αλλά είναι αναγκαιότητα. Βλέπουμε χάο γύρω από τα σύνορά μα, διαλυμένα κράτη, παγωμένε συγκρούσει, στιγνά εγκληματικά συμφέροντα και έμποροι ανθρώπων που κερδοσκοπούν παίζοντα με τη ζωή των ανθρώπων. Ακριβώ για του λόγου αυτού, οι επιχειρήσει του ΝΑΤΟ και τη Frontex στα εξωτερικά σύνορα είναι ορθέ και λαμβάνουν χώρα την κατάλληλη στιγμή. Βοηθούν πραγματικά του ανθρώπου, των οποίων η ζωή κινδυνεύει και αυτό αποτελεί πανανθρώπινη αξία. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να κάνουμε την κατάλληλη διάκριση ανάμεσα σε αυτού που προσπαθούν να σωθούν και στου μετανάστε εκείνου που απλώ αναζητούν δημιουργηθούν καλύτερες οικονομικές προοπτικές. Σήμερα το προσφυγικό ζήτημα είναι κρίσιμη σημασία για την Ευρώπη. Δύναται να αλλάξει την Ευρώπη πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Αναζωπηρώνει δεινά του παρελθόντο όπω ο λαϊκισμό, ο εθνικισμό και οι διχόνοιε. Καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μια καλύτερη κοινή και μακροπρόθεσμη λήψη αποφάσεων. Εν ώψη λοιπόν των πρωτόγνωρων αυτών μεταναστευτικών ροών, κάθε κράτο μέλο πρέπει να καταδείξει αλληλεγγύη και υπευθυνότητα. Η Βουλγαρία έχει αποδείξει ότι είναι ένα πιστό εταίρο και στι καλέ και στι δύσκολε στιγμέ. Βρισκόμαστε στον πιο εύκολο, θα έλεγα και άμεσο δρόμο που ενώνει τι περιοχέ των κρίσεων με τη Δυτική Ευρώπη. Η Βουλγαρία προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο αποτελεσματικό και επαγγελματικό. Ακολουθούμε του κανόνε του Δουβλίνου και του Σέγγεν. Δείχνουμε αλληλεγγύη προ του πρόσφυγε. Χορηγούμε ανθρωπιστικό καθεστώ σε όσου πληρούν τα κριτήρια. Η Βουλγαρία πληρεί όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της ως κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται λοιπόν ισότιμα με τις χώρες του Σέγγεν, με την προσχώρησή της στο χώρο Σέγγεν το συντομότερο δυνατό προς όφελος της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας. Η Βουλγαρία υποστηρίζει τη θέσπιση ενός συστήματος αλληλεγγύης το οποίο θα επιτρέψει δίκαιη μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση των προσφύγων ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προεδρεύων της διαδικασίας συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Βουλγαρία ανέλαβε την πρωτοβουλία για μια κοινή δήλωση για τη μετανάστευση και έθεσε ως θέμα προτεραιότητας για την όλη περιοχή την ασφάλεια και τη μετανάστευση. Σήμερα τα Βαλκάνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία τη Ευρώπη. Θα ήθελα πραγματικά λοιπόν τα Βαλκάνια να γίνουν η πρώτη γραμμή σταθερότητα και ευημερία. Μια πρώτη γραμμή για την ανεκτικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών θρησκειών και εθνοτικών μειονοτήτων. Ω πρόεδρο λοιπόν τη Βουλγαρία λέω το ακόλουθο. Θέλουμε κατάρριψη και όχι μετακίνηση των συνόρων. Έχουμε μια ισορροπημένη εξωτερική πολιτική που διέπεται από αρχέ. Θέλουμε να είμαστε φίλοι με όλου γιατί πιστεύουμε ότι όλοι και ο καθένας μπορούν να συμβάλλουν στην ειρήνη και στη σταθερότητα. Η στενή λοιπόν συνεργασία για τη μετανάστευση και τη μετώπιση της ρίζοσπαστικοποίησης του βίου εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας είναι ένα ακόμη παράδειγμα του ότι πρέπει να συμπορευτούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια. Η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μπορεί να βοηθήσει και τα Δυτικά Βαλκάνια να αφήσουν πίσω τους το βαρύ φορτίο των συγκρούσεων. Εθνικιστικές ιδεολογίες οι οποίες οδήγησαν σε κτηνοδίες ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Συνεπώς η ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας και οι φιλικές ειρηνικές αυτές σχέσεις είναι θεμελιώδου σημασίας για μια πολιτική διεύρυνση και σαφής δείκτης του κατά πόσον οι χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ασπαστεί βασικές ευρωπαϊκές αξίες. Η Βουλγαρία δραματίζει σημαντικό ρόλο προκειμένου να ενισχύσει την εμπειρογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκή Ένωση στην όλη περιοχή. Υποστηρίζουμε στεναρά τη συνεργασία υπέρ μια συμφιλίωση, διασύνδεση και ολοκλήρωση. Η Σύνοδο λοιπόν τη Διαδικασία Συνεργασία για την Νοτιοανατολική Ευρώπη που έλαβε χώρα στη Σόφια την προηγούμενη εβδομάδα τίμησε επίση την 20η επέτειο τη Συνόδου αυτή, η οποία αποτελεί μια αυθεντική φωνή για την όλη περιοχή. Αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει να συνταχθούμε και να αναπτύξουμε κοινέ στρατηγικέ, αντί να οικοδομούμε οχυρά για να προασπίσουμε κοντόφθαλμα εθνικά συμφέροντα. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε ηγέτες ε, από πολιτικούς, οικονομικούς τομείς και τομείς της κοινωνίας των πολιτών. Και ας μην αναλωνόμαστε μόνο σε συζητήσεις, αλλά συμβάλλουμε πραγματικά για να επιλύσουμε τα προβλήματα. Καθώς αναδύονται νέες οικονομικές, δημογραφικές και πολιτικές δυνάμεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις και τους δεσμούς που έχουμε με οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς. Οι Διατλαντικέ λοιπόν σχέσεις είναι στρατηγική σημασία απέναντι σε αυξανόμενε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοκρατική τάξη πραγμάτων. Ένα λαμπρό λοιπόν μέλλον για την Ευρώπη απαιτεί επινόηση ενό νέου οικονομικού μοντέλου. Ενό μοντέλου που θα ανταποκρίνεται σε επερχόμενε προκλήσει και που θα αξιοποιεί το ευρύτατο φάσμα νέων ευκαιριών. Το νέο οικονομικό μοντέλο τη Ευρώπη θα πρέπει να είναι δυναμικό και ανοιχτό. Θα πρέπει να προωθήσουμε νέε προσεγγίσει και μηχανισμού. Α μην φοβόμαστε φαινόμενα όπω η συμμετοχική ή η συνεργατική οικονομία ή όπω το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ανταυτού, α καλωσορίσουμε τα φαινόμενα αυτά και α χρησιμοποιήσουμε όλε τι κοινοτομίε με τον πιο παραγωγικό τρόπο. Η Ευρώπη θα πρέπει να κατακτήσει ηγετική θέση στην νέα βιομηχανική αυτή επανάσταση ηγετική θέση στη λεγόμενη ανατρεπτική οικονομία, ηγετική θέση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Η Ευρώπη του μέλλοντος θα πρέπει να είναι η Ευρώπη των επιχειρηματιών, η Ευρώπη της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Και όντως όλοι θέλουμε μια δυναμική, ευέλικτη, ευπροσάρμοστη Ευρώπη, μια Ευρώπη που να ενώνει και να ηγείται. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Πρέπει να λάβουμε προληπτική δράση. Θα πρέπει να είμαστε προδραστικοί, διορατικοί, να επιλύουμε τις κρίσεις. Θα πρέπει να εστιάσουμε σωστά. Θα πρέπει να επιλέξουμε μια κρίση, να την επιλύσουμε και στη συνέχεια να είμαστε περήφανοι που την επιλύσαμε κατά τρόπο ευρωπαϊκό, με τον δικό μας λοιπόν τρόπο. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε θαραλέες πολιτικές αποφάσεις. Η Ένωσή μας, απεγνωσμένα αυτό χρειάζεται σήμερα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τη διπλωματία, να διαπραγματευόμαστε, να διαπραγματευόμαστε συνεχώς και να μην πολεμούμε, γιατί η χρήση των όπλων αποτελεί απλώ απόδειξη απουσίας επιχειρημάτων. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις αρχές και όχι τα συμφέροντα. Θα πρέπει να εδραιώσουμε εκ νέου και όχι να επαναδιαπραγματευόμαστε τις αρχές του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία, την εδαφική αικαιρεότητα, την κυριαρχία και να προσπιζόμαστε επίσης το παραβίαστο των συνόρων κάθε κράτους μέλου στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ναι, έχουμε μπροστά μας αυξανόμενους κινδύνους και αυξανόμενη αβεβαιότητα, καθώς κινούμαστε προς μια πιο ασταθή παγκόσμια τάξη και νόντως θα απαιτηθεί χρόνος προκειμένου να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια νέα ισορροπία, σε έναν νέο πολυπολικό κόσμο. Σε αυτή τη μεταβατική λοιπόν περίοδο θα πρέπει να οικοδομήσουμε και να επανοικοδομήσουμε μια πιο ανθεκτική περιφερειακή και παγκόσμια τάξη μέσω των δικών μας κοινών προσπαθειών. Θα πρέπει να προωθήσουμε θεσμικές μεταρρυθμίσεις, διπλωματία και αρχές. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους ηγέτες εκείνους οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύονται ειρηνικά και όχι μέσω πολέμων διαντιπροσώπων ή προπαγανδιστικών πολέμων. Και θα πρέπει να δείξουμε στεναρή στάση, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε απλώς θα ενθαρρύνουμε τους ανεύθυνους εκείνους ηγέτες οι οποίοι επιθυμούν να αποσταθεροποιούν όλο και περισσότερο. Αγαπητοί φίλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί καθημερινή επιβεβαίωση της επιθυμίας μας να ζούμε μαζί. Η ιστορία καταδεικνύει ότι χωρίς συνεχείς προσπάθειες οτιδήποτε έχουμε κερδίσει μπορεί να χαθεί. Οι συζήτηση που γίνονται για την μετανάστευση, για το Brexit, οι λαϊκιστέ, οι ευρωσκεπτικιστέ επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα αυτό σήμερα περισσότερο από ποτέ. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο κοινό μα ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο είναι ζωτική σημασία και για το οποίο δεν υπάρχει εναλλακτική. Θα πρέπει να διασκεδάσουμε του φόβου των Ευρωπαίων και να του διασφαλίσουμε ότι ξέρουμε πραγματικά προ τα που οδεύουμε. Η σημερινή Ευρώπη οδηγεί σε περισσότερε ερωτήσει και λιγότερε απαντήσει. Οι πολίτε μα χρειάζονται περισσότερη ασφάλεια σε έναν όλο και λιγότερο ασφαλή κόσμο και διαρωτώνται πώ μπορούμε να ζήσουμε αρμονικά με του γειτονέ μα. Η ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και ευθυνών στην ευρωπαϊκή κοινωνία αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρο τη απάντηση που πρέπει να δώσουμε. Θα πρέπει να δείξουμε προ τον έξω κόσμο αλλά και προ του πολίτε μα ότι όντω έχουμε εμπιστοσύνη στι δυνατότητέ μα και ότι μπορούμε μάλιστα να τι ενισχύσουμε. Θέματα όπω η μετανάστευση, η τρομοκρατία, οι παγωμένε συγκρούσει δεν μπορούν να επιληθούν αν δεν αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια. Γεωπολιτικά αποθυμένα και διαχρονικέ βαθιά ριζωμένε συγκρούσει. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση των κρίσεων και μπορούμε να σχεδιάσουμε και την επίλυση των κρίσεων αυτών από στρατηγική πλευρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είμαστε ρεαλιστέ. Τα περισσότερα προβλήματα έχουν κοινωνικά ε, ευρωπαϊκά αίτια, κοινωνικός αποκλεισμός, περιθωριοποίηση, ανεπαρκής παιδεία, ανεπαρκής διάλογος μεταξύ των θρησκειών. Και γι' αυτό τον λόγο οδηγούμαστε σε ρίζος παστικοποίηση. Η τρομοκρατία ξεκινάει εκεί πέρα που αποτυχαίνει η παιδεία και η εκπαίδευση. Πολλοί τρομοκράτες και αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές είναι Ευρωπαίοι. Α μην ξεχνάμε την ηθική μα υποχρέωση να αποτελέσουμε χώρο ελευθερία και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όσου κινδυνεύουν είναι θύματα καταδυνάστευση. Αλλά επίση ε, προασπίζουμε κανόνε και αξίε που αντιστοιχούν συγκεκριμένα δικαιώματα και ευθύνε. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η εκπαίδευση, η κοινωνική ενσωμάτωση αποτελούν δέσμευση τόσο για τι κοινωνίε υποδοχή όσο και για του πρόσφυγε. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι προφανέ ότι χωρί βασικέ πολιτικέ και λύσει, οι οποίε θα προκύπτουν από τον διάλογο, οι φόβοι των πολιτών θα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από του λαϊκιστέ. Χωρί μια ρεαλιστική προσέγγιση θα είναι δύσκολο να απορρίψουμε τι εικασίε αυτέ που λένε ότι ορισμένοι επιθυμούν να οικοδομήσουμε την Ευρώπη κρυφά από του Ευρωπαίου πολίτε. Οι λαϊκιστέ και οι εθνικιστές μας, αναγκάζουμε, μας αναγκάζουν να επιλέξουμε ανάμεσα στις αρχές που κληρονομήσαμε από τους ιδρυτές της Ένωσης και την ανάγκη να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πολιτών. Εμείς επιλέγουμε και τα δύο. Επιλέγουμε και τις αξίες και την ασφάλεια. Και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει καμία αντίφαση ανάμεσα στο να προασπίζουμε τα σύνορά μας και από την άλλη να τηρούμε τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Και βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους εθνικιστές και τους πατριώτες. Ένας σπουδαίος Ευρωπαίος πρόεδρος, ο πρόεδρος Ντεγκόλ, είχε πει κάποτε «Οι πατριώτες είναι αυτοί που αγαπούν τη χώρα τους. Οι εθνικιστές είναι αυτοί που μισούν οτιδήποτε το διαφορετικό». Σήμερα λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, Σήμερα λοιπόν περισσότερο από ποτέ Χρειαζόμαστε έναν σύγχρονο πατριωτισμό και όχι έναν επιθετικό εθνικισμό στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, οι κοινέ αρχές και η σφαιρική προσέγγιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθοριστική σημασία για το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Είναι σαφές ότι οι εθνικές κοινωνίες διαφέρουν μεταξύ τους και έχουν διαφορετικές αντιδράσεις από ιστορικής πλευρά σε διάφορα γεγονότα αλλά στη διαφορετικότητα αυτή τη ιστορία και του πολιτισμού μα βρίσκεται το πλούτο τη Ευρώπη. Αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει όμω λόγο για να τροποποιήσουμε τη φύση του ευρωπαϊκού σχεδίου, δημιουργώντα μια Ευρώπη δύο περισσότερων ταχυτήτων. Η ισότητα της ευρωπαϊκής δέσμευσης λοιπόν έχει άμεσες συνέπειες στην ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Ακόμα και η υπόνοια, η υπόνοια και μόνο ότι μπορούμε να αποδεχτούμε μια Ευρώπη διαφορετικών ταχυτήτων στέλνει από μόνο του ένα μήνυμα αμφισβήτησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπονοεί τελικά μια ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήταν πραγματικό σφάλμα να υποτιμήσουμε την δυνατότητα ανάπτυξη ορισμένων περιοχών τη Ευρώπη. Να υποτιμήσουμε, για παράδειγμα, τα Βαλκάνια. Θα ήταν ιστορικό σφάλμα να μην υποστηρίξουμε τα Βαλκάνια ή να τα αφήσουμε έρμεο στην επιρροή ξένων δυνάμεων. Δεν θα πρέπει να στρέφουμε τα ευρωπαϊκά έθνη του ένα εναντίον του άλλου. Μόνο μία απάντηση μπορεί να δοθεί αλληλεγγύη προς τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν μπροστά τους, ιδίως σε μια περίοδο προκλήσεων και αντικσοτήτων. Η αλληλεγγύη αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει τα απλά μέσα της πολιτικής συνοχής και να αποτελεί τμήμα οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πολιτικής. Ανεξάρτητα από την έκβαση του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασίλειο, η συζήτηση για την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα συνεχιστεί. Θα πρέπει να αποφύγουμε την καταστρεφική αυτή φύση της όλης συζήτησης της Ευρώπης Αλακάρτ. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε Έχουμε μόνο όποτε μας αρέσει την αλληλεγγύη και να κάνουμε τελικά την Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς ένα σύνολο συναλλαγών και δοσοληψιών. Και αυτό διότι κάθε χώρα έχει διαφορετικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Επομένω, αυτό το παιχνίδι μηδενικού αθρίσματος έχει και είχε και στο παρελθόν καταστροφικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να φουγκραστούμε καλύτερα τους εταίρους μας. Η Βουλγαρία αποτελεί ένα παράδειγμα μιας χώρας μεσαίου μεγέθους που από περιφερειακή χώρα έγινε χώρα πρώτης γραμμής. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη μετανάστευση. Τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Οι γειτονές μας είναι σύνορε είναι γείτονε, με τη Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε δύσκολε επιλογέ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σκεφτήκαμε να θυσιάσουμε την ευρωπαϊκή ελληνική. Διότι εμεί, οι Βούλγαροι, έχουμε μάθει πλέον ότι δεν μπορούμε να αλλάζουμε τη γεωγραφία. Και ότι η πραγματική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορεί τελικά να βρει ευκαιρίες στα πλαίσια των γεω... γεωγραφικών κινδύνων. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωπαϊκέ δημοκρατίε δεν είναι τέλειε και δικαιολογημένα πολλέ φορέ δέχονται επικρίσει. Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε πολύ καλύτεροι από άλλου. Δεν μπορούμε να πείσουμε του ευρωσκεπτικιστέ, αλλά θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τουλάχιστον του Ευρωπαίου. Θέλω να το καταστήσω σαφέ. Όλες αυτές οι προβλέψει για την αποτυχία και την αποσύνθεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λανθασμένε και ψευδείς. Έχουμε αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις στην ιστορία μας. Και η θεραπεία είναι σαφής. Περισσότερη ελεγγύη, περισσότερη ανθρωπιά, περισσότερη συμπόνια, περισσότερο κράτος δικαίου, περισσότερη συνεργασία, περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη ολοκλήρωση. Ο πρώτος δημοκρατικά κλεγμένος βούλγαρος πρόεδρος, Ζέλιου Ζέλεφ, έλεγε Μπορεί να θεραπεύσει κανεί τη δημοκρατία μόνο με περισσότερη δημοκρατία. Είμαι πεπισμένο λοιπόν ότι θα αντιμετωπίσουμε όλε αυτέ τι προκλήσει χωρί να υπονομεύσουμε τι βασικέ μα αξίε. Το έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό στο παρελθόν και θα ήταν πραγματικό λάθος αν ορισμένοι ερμηνεύουν την ανεκτικότητά μας ως αδυναμία. Αντίθετα, αποτελεί σήμα αποφασιστικότητας δύναμης, ότι εμείς θέλουμε να καθορίσουμε τη ζωή μας. Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας έχει διδάξει ότι σε περιόδους αντικσότητας μόνο η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση λειτουργεί. Το μόνο όπλο που έχουμε στα χέρια μας για να πετύχουμε την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανθρώπινη ανάπτυξη είναι η ολοκλήρωση. Μια χώρα από μόνη της δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Τον αρθώνουμε σύνορα. Ακόμα και αν είναι αυτά εδαφικά, οικονομικά ή νομικά είναι μια δελεαστική αλλά ουσιαστικά προσωρινή και μη βιώσιμη λύση. Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ σοβαρές και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δεν μπορούμε να μεταθέτουμε τα προβλήματα στην επόμενη κυβέρνηση, στην επόμενη γενιά. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση, να αναλάβουμε, να λάβουμε αποφάσεις το μότρο δυνατό. Δεν έχουμε την επιλογή της αδιαφορίας αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να γνωρίζουμε πώς θα τα επιλύσουμε. Υφίστανται πολλές κρίσεις. Μία από αυτές είναι ότι σήμερα η Ρωσία δεν υποστηρίζει τις αρχές της διεθνούς τάξης. Το Κρεμλίνο αντιτίθεται πλέον σε εμά και προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφυσώντα δυσπιστία στην ίδια την καρδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματο. Προσπαθεί να καταστρέψει και να καταρρύψει τα ίδια τα θεμέλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είναι η ενότητα, η αλληλεγγύη και το κράτο δικαίου. Η άρχισε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση προπαγάνδας στην Ευρώπη με στόχο να διασπείρει μηνύματα δυσπιστίας και όχι συγκεκριμένες αρχές. Στόχος να απονομευτεί η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερο κίνδυνος, θα έλεγα. Το να διαβρωθεί η εμπιστοσύνη των ίδιων των Ευρωπαίων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και στο κοινό μας πεπρωμένο. Το να επιστρέψουμε τελικά τον επιτρέψουμε στα φαντάσματα του παρελθόντος να επιστρέψουν. Εθνικισμός, λαϊκισμός, μεγάλες δυνάμεις, σφαίρες επιρροής, συμφέροντα, όλοι αυτοί οι παράγοντες που ουσιαστικά στρέφονται κατά των αρχών και των αξιών. Και από ό,τι φαίνεται η Ρωσία σημειώνει πρόοδο. Εμείς από την άλλη δεν σημειώνουμε πρόοδο. Έχουμε σταματήσει τη βασική κινητήρια δύναμή μας, την ολοκλήρωση. Επιβραδύνουμε αυτή τη στιγμή το Σέγγεν και τη διαδικασία διεύρυνσης θεωρώ ότι θα πρέπει να ανοίξουμε διάπλατα τις πόρτες ανταυτού, να ατενίσουμε νέους ορίζοντες. Θα πρέπει να βάλουμε πάλι μπρο τη μηχανή αυτή τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, να ξεκινήσουμε νέα σχέδια ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε και να ενισχύσουμε τα θεμέλια τη τάξη και των αρχών μα, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούμε επίση και σε έναν κόσμο ο οποίο μεταλλάσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να ενσωματώνουμε και να μην απομονώνουμε. Θα πρέπει να κοιτάμε μπροστά και όχι πίσω. Η Ευρώπη μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό παγκόσμιο ρόλο και θα πρέπει να κινητοποιηθεί, να ξεκινήσει νέα προγράμματα ολοκλήρωσης και θα πρέπει να δούμε και την δοπιό διαφορά ανάμεσα στην τεχνική αντιμετώπιση των πραγμάτων και το περιεχόμενο. Το μέλλον της Ευρώπης δεν έχει να κάνει με την τεχνική φύση των πραγμάτων. Τα μία για το ευρώ, οδηγίε, διαχείριση των κρίσεων και όλα αυτά. Το μέλλον τη Ευρώπη ανταυτού έχει να κάνει με το πραγματικό περιεχόμενο του οράματός μας. Τι πραγματικά θέλουμε και ποιοι είμαστε. Ουσιαστικά βασική αρχή είναι το κράτο δικαίου. Το μέλλον τη Ευρώπη έχει να κάνει με το να μην ξεχνάμε τις σημαντικές ιδέες. Δεν θα πρέπει απλώς να επικεντρωνόμαστε στις τεχνικές λεπτομέρειες. Ας μην χάνουμε τη σφαιρική εικόνα. Ας δούμε πραγματικά ποιο είναι το όραμά μας για την Ευρώπη. Πώς προσδίδουμε προς τη θέμενη αξία στην εργασία που έχουν κάνει οι προηγούμενες γενιές πώς προσδίδουμε προς τη θέμενη αξία στο όραμα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρωτώ με πώς σκέφτονταν οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είχαν κατά νου πριν από 70 χρόνια μετά την καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ε, όλοι μισούσαν τους πάντες στην Ευρώπη. Γνώριζαν τότε οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η ειρήνη μπορεί να επικρατήσει μόνο όταν τα έθνη έχουν τέτοιο βαθμό συνεργασίας που οποιοδήποτε πόλεμο στο μέλλον είναι αδύνατος. Και έτσι ξεκίνησαν τη διαδικασία της ένωσης και της ε, ολοκλήρωσης στο χάλιβα, στον άνθρακα και σε άλλους τομείς. Η βασική ιδέα δεν ήταν να αποδυναμώσουν τα εθνικά κράτη, αλλά να τα καταστήσουν ισχυρότερα μέσω της ένωσης. Η Βουλγαρία ήταν πάντα δύναμη όσο ήταν μόνη της. Η Βουλγαρία είναι ισχυρή σήμερα ως περήφανο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή είναι πού θέλουμε να φτάσουμε το 2030, το 2050. Προφανώ θα πρέπει να λύσουμε το ζήτημα τη μετανάστευση, την τραπεζική κρίση, το χρέο και τι υπόλοιπε χρήσει, αλλά θέλουμε πραγματικά να περιοριστούμε σε αυτά. Θέλουμε να κάνουμε μόνο διαχείριση κρίσεων πηγαίνοντα απλώ από τη μία κρίση στην άλλη. Μα αυτό ουσιαστικά είναι μόνο τεχνοκρατική προσέγγιση. Δεν συνιστά όνειρο ούτε όραμα. Εγώ θέλω να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία όπω και ιδρυτέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να βάλουμε πάλι μπρο τι μηχανέ τη ολοκλήρωση, τη διαδικασία τη διεύρυνση, για παράδειγμα. Μια πιο αποτελεσματική και συντονισμένη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Μια ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση. Μια ενιαία ψηφιακή αγορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ευρωπαϊκή ένωση κεφαλαγορών. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να διαμορφώνουμε και να γράφουμε την ιστορία, μια ιστορία μιας, ευρωπαϊκής, μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης με δυνατά και βήμαρα κράτη. Αν ξεχαστούμε και δεν έχουμε πλέον στόχους, κάποιος θα επικεντρωθεί εκ νέου σε εμά και θα μας θεωρήσει βολικό και εύκολο εχθρό. Αν σταματήσουμε να γράφουμε ιστορία, κάποιος άλλος θα τη γράψει για μας. Καθώς ορισμένοι αμφισβητούν και θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τις βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταυτού εμείς ας ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας το πράξουμε τώρα όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τον πολύ θαραλέο λόγο σας. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τη συμμετοχή σας μέσω των εντόνων χειροκροτημάτων. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπα, είναι ιδιαίτερα τολμηρός ο λόγος σας. Και από τις αντιδράσεις ε, διαπιστώνεται ότι στην πληθυντική πλειοψηφία των συναδέλφων συμμερίζονται την άποψή σας, αλλά σίγουρα υπάρχουν και συνάδελφοι στο σώμα που έχουν εντελώς διαφορετική άποψη και πρέπει να πω ότι εγώ ανήκω στην πρώτη ομάδα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το θαραλέο λόγο σας. Σας ευχαριστώ.